Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση του κυρίου Λέχνα ε, με θέμα κληρονομική διαδοχή και ευρωπαϊκό κληρονομητήριο. Ο εισηγητής, ο κύριος Κουρτ Λέχνα, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρία επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι, για το τον Ευρωπαίο πολίτη ο οποίος έχει περιουσιακά στοιχεία ε, σε μία άλλη χώρα είναι πολύ δύσκολο να οργανώσει τη διαδοχή του. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία είναι άλυτα και κοστίζουν πάρα πολλά χρήματα. 12 εκατομμύρια υπήκοοι της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ζουν σε μία άλλη χώρα και πολλοί από αυτούς έχουν ποεριουσία και υπάρχουν επιπλέον άλλα τρία εκατομμύρια τουλάχιστον υπήκοοι άλλων χωρών που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτοί πλήγονται από όλα αυτά τα προβλήματα. Αυτή τη στιγμή μπορεί ο πολίτης να καθορίσει ποιος θα τον κληρονομήσει. Αλλά εάν δεν υπάρχει διαθήκη τότε ε, θα πρέπει ε, να ξεκινήσει η ρύθμιση των περιουσιακών του στοιχείων από τη χώρα όπου διέμενε αλλά πρέπει να αποδείξει ε, που υπήρχε η κυρία έδρα του να μην υπάρχει πλέον δηλαδή αμφιβολία επ' αυτού. Εν αντιθέσει με την μέχρι τώρα κατάσταση Τώρα θα υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση και οι κληρονόμοι οι οποίοι μπορεί να μάχονταν σε πολλά κράτη με τα δικαστήρια τώρα θα μπορούν να απευθύνονται σε ένα διεθνές χώρο όπου θα υπάρχει ένα μητρό και ε, θα μπορεί να ρυθμίζει τα θέματα του κληρονομητηρίου πράγμα το οποίο θα απλοποιήσει τη διαδικασία και θα εξοικονομήσει και χρόνο και χρήματα. Θα ήθελα να σας ε, αναφέρω ορισμένα σημεία. Εδώ δεν μιλάμε για την φορολογία κληρονομίας διότι αυτή δεν αλλάζει αλλά θα ακολουθήσει την πρώτη δεύτερη ερώτηση την οποία θέτουν οι, περί, πολίτες. Δεύτερον το δίκαιο της κληρονομίας δεν αλλάζει αλλάζει. Οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν τρία χρόνια μετά από την εφαρμογή της ρυθμίσεως και τέταρτον για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία ισχύει ένα opt-out το οποίο ίσως καλύψει και την Δανία. Ελπίζουμε όμως ότι ε, δεν ε, θα υπάρξει μία κωδικοποίηση των μέχρι τούδε υπαρχόντων συνθήκων αλλά μία δημιουργία ενός νέου δικαίου και η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ιδιαίτερα καλή και πρέπει να το αναγνωρίσουμε και να το χαιρετήσουμε. Επίσης επί δυόμιση χρόνια υπάρχει συζήτηση που οδήγησε σε, πολύ καλή, σε πολλές βελτιώσεις και εδώ χαιρετίζω τη συνδρομή των συναδέλφων της νομικής επιτροπής οι οποίοι μπόρεσαν να βελτιώσουν πολύ το κείμενο αλλά το ίδιο ισχύει και για το Συμβούλιο γιατί έχει επεξεργαστεί πάρα πολύ ενδελεχώς την πρόταση αυτή και μπόρεσε να τη βελτιώσει. Ιδιαιτέρως ευχαριστώ την Δανική Προεδρία η οποία μπόρεσε να βελτιώσει ακόμη περισσότερο την πρόταση. Επίσης η συζήτηση συζητήσεις διεξήχθησαν πάρα πολύ θετικά. Γι' αυτό, κυρία Επίτροπε, επειδή ακριβώς είδατε ότι μιλούσαμε για την ισοτιμία των φύλων, να σας πω ότι εδώ ουσιαστικά πρέπει να σας πω ότι οι βελτιώσεις ε, επήλθαν από γυναίκες τις οποίες χαιρετίζω. Ε, τώρα θα είναι πολύ απλοποιημένη η διαδικασία παρόλο που έπρεπε να απαντήσουμε σε πολύ δύσκολα ερωτήματα. Όλα μπόρεσαν να, να επιληθούν προς όφελος των πολιτών κατά τρόπον όλοι να μπορέσουν να αποδώσουν. Σας ευχαριστώ. Τώρα το λόγο έχει εξ ονόματος της Επιτροπής η Αντιπρόεδρος κυρία Ρέντιν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που βλέπω ότι είναι στην ημερήσια διάταξη αυτής της Ολομέλειας η... το θέμα αυτό διότι οι πολίτες της Ευρώπης περιμένουν για υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα. Το Συμβούλιο το 2000 επεσήμανε αυτό το πρόβλημα σαν, τομέας για δράση, σαν τομέα για δράση. Και είναι πρώτη φορά που θεσπίζεται ένα ευρωπαϊκό μέσο στον τομέα των κληρονομιών. 10% περίπου του συνολικού αριθμού διαδοχών και κληρονομιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν μια διεθνή διάσταση. Μιλάμε για 120 δισεκατομμύρια ευρώ αξία. Ο κανονισμός λοιπόν αυτός αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να δείξουμε ότι η Ευρώπη αποφάσισε να ενεργήσει για να καταστήσει πιο εύκολη τη ζωή των πολιτών που βρίσκονται αντιμέτωποι με περίπλοκες νομικές καταστάσεις. Γνωρίζω πολύ καλά ότι το θέμα των κληρονομιών είναι ένα θέμα ευαίσθητο που συνδέεται με τις εθνικές πολιτικές για την προστασία της οικογένειας και εθνικά ε, νομικά συστήματα και υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές ανάμεσα στην εθνική συνενομοθεσία των διαφόρων χωρών. Ευτυχώς έχουμε όμως έναν θαυμάσιο εισηγητή, τον κύριο Λέχνερ θα είναι μια από τις τελευταίες ενέργειες που έχει αναλάβει σε αυτό το κοινοβούλιο από ό,τι αντιλαμβάνομαι διότι θα αποσυρθεί. Με, αυτό, με αυτή τη δράση έχετε αφήσει μια σφραγίδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κύριε Λέχνερ και όλοι πρέπει να σας ευχαριστήσουμε για τις προσπάθειες που κάνατε για το καλό προς των πολιτών της Ευρώπης τα αποτελέσματα που προτείνει ο εισηγητής είναι εντυπωσιακά και η Επιτροπή θα υποστηρίζει απόλυτα και το ψήφισμα που ε, θα εγκριθεί αύριο επιτηρεί τους σωστούς στόχους που είναι ε, ε, για την Επιτροπή το εξή ότι θα υπάρχει ένας, ένα, ένα, θα ισχύει μόνο ένας νόμος στο, χώρα, στον τόπο κατοικίας οι πολίτες θα έχουν την ελευθερία να διαλέξουν τη χώρα της, της του τους ανάλογα με το πώ μετακινούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα υπάρχει ελεύθερη κυκλοφορία των δικαστικών αποφάσεων στην Ευρώπη. Και βεβαίω το κερασάκι στην τούρτα είναι το Ευρωπαϊκό Κληρονομητήριο που θα επιτρέπει στους, στα άτομα να ασκούν τα δικαιώματά τους ως κληρονόμων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνώ απόλυτα με τον εισηγητή. Το κείμενο που συζητούμε ε, εδώ και πάρα πολύ καιρό έχει βελτιωθεί ουσιαστικά χάρη στις σκληρές προσπάθειες του εισηγητή και της Επιτροπής επιμένοντας στην εξασφάλιση νομικής βεβαιότητας για εκείνους οι οποίοι χρειάστηκε να κάνουν ορισμένα πράγματα προτού περάσει αυτό το κείμενο. Σας συγχαίρουμε και πάλι. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα θέματα που μπορούμε να φέρουμε στο τραπέζι στη διάρκεια αυτού του έτους, δείχνοντας έτσι ότι πραγματικά φροντίζουμε και μεριμνούν για τους πολίτες. Πρόεδρο της Κομισιόν, τώρα το λόγο έχουν οι ομιλητές εξ των πολιτικών ομάδων. Δίνω το λόγο στον κύριο, στον κύριο Κλάους Χάινα Λένε, εξ ονόματος της κοινοβουλευτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος των Χριστιανοδημοκρατών. Κύριε Λένε, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμε κύριε Σιγητά, κυρία Επίτροπε, είναι ουσιαστικά κρίμα διότι δεν μαθαίνουμε ποτέ. Είναι νύχτα, συζητάμε ένα πολύ σημαντικό νομοθέτημα το οποίο όπως είπε η Επίτροπος αφορά 10% των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, δηλαδή 50 εκατομμύρια κατοίκου οι οποίοι είτε άμεσα είτε έμεσα πλήττονται και λόγω των ε, συνθήκων είναι νύχτα, δεν είναι και τόσοι πολλοί, ίσως η διάσκεψη των ε, προέδρων ε, δεν θα μπορούσε να σκεφτεί να μεταφέρουμε μία ανούσια συζήτηση για μία διάσκεψη κορυφής και να γίνει μία τέτοια σημαντική συζήτηση κάποια ώρα όπου υπάρχουν ε, περισσότεροι παριστάμενοι διότι είναι κάτι πολύ βασικό και είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο δηλαδή είναι ένα πολύ περίπλοκο θέμα και θέλω αυτό να το τονίσω διότι σαν ε, επικεφανής της νομικής επιτροπής ε, θέλω να χαιρετήσω τον κύριο Λέχνερ ο οποίος είναι ένα από τα πιο ικανά μέλη του Κοινοβουλίου και να του πω ότι ουσιαστικά αυτό ήταν το χαιρετιστήριό του δώρο που είναι πολύ πολύτιμο διότι είναι ένα αξιόλογο δώρο από χαιρετιστήριο και το τονίζω διότι όπως μας είπε στο τέλος της εβδομάδος θα μας αποχαιρετήσει, θα καταθέσει την εντολή του και θέλω να του πω και πάλι ότι λυπούμε πάρα πολύ ότι μας εγκαταλείπει διότι αυτό το οποίο αποφάσισε το Συμβούλιο ε, δείχνει ότι το Συμβούλιο απλώς εάν ακολουθούσε την πρόταση Λέχνερ θα είχαμε ένα ολοκληρωμένο φάκελο που θα βοηθούσε τους πολίτες να μπορέσουν να διεκπαιρεώσουν τα θέματά τους και να προωθήσουμε την Ευρώπη των πολιτών. Σας ευχαριστώ. Ο ομιλητής είναι ο κύριος Λουίτζι Μπερλιγκουέρ, εξ της ομάδας της των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κύριε Λουίτζι ε, Μπερλιγκουέρα, έχετε το λόγο για τρία λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, καταρχήν. Και εγώ θα ήθελα να αποτείνω έναν θερμό χαιρετισμό προς τον κύριο Λένε για την εξαιρετική του εργασία, στην οποία ανταποκρίθηκε με αποφασιστικότητα. Πολλές φορές ε, είχαμε ε, προσκρούσει σε εμπόδια, αλλά πάντα τα κατάφερνε να ανταποκριθεί. Και νομίζω ότι είμαστε ομόφωνοι ως προς αυτό. Τώρα, ως προς τον κανονισμό κάθε αυτό, είμαι πεπισμένος ότι είναι κάτι το σημαντικό. Ίσως ε, δεν έχει απήχηση στον τύπο, δεν θεωρείται υψηλή πολιτική, αλλά η οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης περνά και από την ικανοποίηση των ε, συμφερόντων, των ενδιαφερόντων και των μελημάτων των ε, πολιτών στην καθημερινή του ζωή. Δηλαδή να υπάρχει μία ανταπόκριση στην καθημερινή του ζωή των ε, πολιτικών που ορίζουμε. διότι έχουμε να κάνουμε με ευαίσθητα ζητήματα, έχουν να κάνουν με τον πυρήνα της οικογένειας. Είμαστε υπερήφανοι διότι καταφέραμε να ανταποκριθούμε. Οι λύσεις είναι ευφυείς και νέες, καινοτόμες, δηλαδή μέσα στα πλαίσια του κληρονομητηρίου μπορεί κανείς να επιλέξει ή την χώρα προέλευσης ή την χώρα κατοικίας. Αυτό δείχνει μία ευελιξία γιατί πολλές φορές μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει προβλήματα εάν δεν γίνεται αυτός ο διαχωρισμός. Και όταν βρούμε την νομική βάση, χώρα προέλευσης ή χώρα κατοικίας, τότε υπάρχει ένας περιορισμός της διακριτικότητας, της διακριτικής ευχέρειας των δικαστών. Υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία και μεγαλύτερη ασφάλεια και ως προς το κληρονομητήριο Θεωρούμε ότι δεν έχει και τόση σημασία, έχει όμως και πολύ μεγάλη μάλιστα, διότι ο κληρονόμος μπορεί να δράσει πιο ελεύθερα με βάση τις ενδεχόμενες δυσκολίες που ανακύπτουν. Βεβαίως ο νόμος δεν είναι τέλειος. Υπάρχουν ε, θέματα εκτέλεσης και ούτω καθεξής. Θα ήθελα μόνο το εξής να πω, ότι ελπίζω το Συμβούλιο να μετατραπεί σε κανονισμό, όχι όμως να ε, θάψουμε αυτό το κείμενο. Δεν θα πρέπει να μην λάβει υπόψη και το Ηνωμένο Βασίλειο τις δυσκολίες που υπάρχουν για να τις υπερβούμε. Δίνω τώρα το λόγο στην κυρία Αλεξάνδρα Τάιν, εξ ονόμα της ομάδας Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, για δύο, για λεπτά. Κυρία Επίτροπε, αξιότιμες κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να προσαρμόσουμε το κληρονομικό δίκαιο και ε, να το αναμορφώσουμε σχετικά με το χώρο κατοικίας και αύριο θα υπάρξει ψηφοφορία. Οπότε σήμερα δεν προσπαθούμε να ρυθμίσουμε αφηρημένες ε, έννοιες αλλά ουσιαστικά διάφορα προβλήματα τα οποία είχαν παραμείνει άλυτα διότι πολλές φορές σε διασυνοριακές κληρονομίες ενδέχεται να υπάρχουν ενδιαφερόμενοι οι οποίοι καταφεύγουν στα δικαστήρια διαφόρων χωρών και συνεχίζουν την νομική διαμάχη επί χρόνια πράγμα το οποίο προσπαθούμε να αποφύγουμε διότι τώρα για το θέμα της εγκατάστασης και το θέμα της διαδοχής υπάρχει μια συγκεκριμένη ρύθμιση και ε, πρέπει αυτή η ρύθμιση να έχει σχέση με το χώρο διαμονής. Αλλά εάν κάποιος που μένει στο Στρασβούργο πιστεύει ότι έχει στενότερες σχέσεις με τη Γερμανία μπορεί να επιλέξει το γερμανικό δίκαιο και αν δεν ε, θέλει το γαλλικό δικαστήριο να χρησιμοποιήσει περίπλοκη γερμανική νομολογία μπορεί να υπάρξει ρύθμιση του θέρματος στα γερμανικά δικαστήρια και η ε, φορολογία δεν πλήττεται από αυτό και από ό,τι ακούσαμε ότι βάσει του οπτά ότι η ε, Βρετανία, η Ιρλανδία και η Δανία δεν θα ακολουθήσουν και είναι κρίμας διότι αυτά δεν θα ακολουθήσουν πλέον το δικαίωμα, το δίκαιο της διαμονής του θανόντος και θα πρέπει να βρεθεί μία λύση πρέπει όμως να ευχαριστήσουμε τον κύριο Λέχνερ ο οποίος δεν ήταν μόνο επαγγελματίας πολιτικός αλλά επαγγελματίας πρακτικός του χώρου για το έργο του. Ευχαριστώ. Λίχτεμπεργα, εξ ονόμα της ομάδας των Πρασίνων της Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να, ξεκινήσω την ομιλία μου ευχαριστώ τον συνάδελφο Λέχνερ ο οποίος έκανε εξαιρετική εργασία και τους σκιώδεις εισηγητές τους οποίους εισάκουσε. Η τωρινή απόφαση προσαρμόζεται εις το κληρονομικό δίκαιο βάσει των εξελίξεων διότι οι άνθρωποι κινούνται, ζουν έξω από την χώρα προελεύσεώ τους και όταν υπάρχουν υπάρχουν κληρονομικά θέματα θα πρέπει κληρονόμοι τους να μπορούν να αποφθυνθούν ε, ενδεχομένως στο κράτος προελεύσεως το οποίο μπορεί να δημιουργήσει πολλές περιπλοκές. Άρα καλό είναι που ελήφθη τώρα αυτή η απόφαση παρόλο που ακόμη μία φορά η πολλαπλή φορά η, η Μεγάλη Βρετανία δεν θα ακολουθήσει. Ε, η χώρα αυτή σε πολλά δεν συμμετέχει αλλά αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι ότι σε περίπτωση ε, ζεύγων ιδίου φύλου δεν θα υπάρχει διάκριση όταν ε, πρόκειται για τα κληρονομικά δικαιώματα τα οποία ε, θα πρέπει να μπορέσουν να ρυθμιστούν βάσει με την επιλογή τους για το κληρονομητήριο και έτσι βλέπουμε βλέπουμε ότι τα πράγματα άλλαξαν και είμαστε σε μια νέα εποχή. Ευχαριστώ. Κύριο ε, Σατζάτ Καρίμ, για δύο λεπτά εξ ονόματος της ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών. Thank you. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι που θα ε, στρέφονται, στρέφονται εναντίον μου διότι αναφερόμενοι στη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον συνάδελφο Λέχνερ για τις τεράστιες προσπάθειες που κατέβαλε για να ετοιμάσει αυτό το κείμενο στη, σε διάρκεια δύο ετών. Τον συγχαίρω και τον ευχαριστώ για όλες τις προσπάθειές του. Έχει συμβάλει, έχει συμβάλει ουσιαστικά και του εύχομαι κάθε καλό όταν ε, θα αποχωρήσει. Θα μας λείψει πολύ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη χρονική συγκυρία, η συζήτηση αυτή είναι σημαντική. Πρόκειτο να συναντηθώ με τον κύριο Λένικτον του Ηνωμένου Βασιλείου, ε, ε, Άγγλου Υπουργού, σήμερα το βράδυ και θέλω να εκφράσω την απογοήτευσή μου διότι που βρέθηκαν το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία σε μια κατάσταση όπου δεν είχαν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν αυτό τον κανονισμό. Έχω πει ότι οι πρακτικές επιπτώσεις θα παραμείνουν και θα είναι αληθινές και θα επηρεάσουν σημαντικά τη ζωή πολλών Ευρωπαίων πολιτών. 50% των κληρονομιών και στο Ηνωμένο Βασίλειο είχαν διασυνοριακό στοιχείο. Μεγάλο ποσοστό, ποσοστό των κατοίκων του Ηνωμένου Βασιλείου προέρχονται από άλλο κράτος μέλος. Οπότε άτομα που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία και θα επηρεαστούν οπωσδήποτε από, αυτό, από αυτό το, τον κανονισμό. Υπάρχουν διατάξεις στον κανονισμό που αφορούν διοικητικά θέματα. Πρέπει να σκεφτούμε κατά πόσο το τελευταίο άρθρο θα καλύψει τις ανάγκες των κατοίκων όλων των κρατών μελών. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι η δεύτερη ανάγνωση κύριε Πρόεδρε, έστω και σύντομη, θα μας δώσει λίγο κάποιο περιθώριο να ξανασκεφθούμε, να ξανασκεφθούμε με πιο φρέσκο μυαλό τα, τα προβλήματα και τις δυσκολίες που ενδεχομένως θα υπάρξουν, ώστε να τις ξεπεράσουμε με, με μεγαλύτερη ευκολία. Ευχαριστώ. Είναι ο κύριος Γιάροσλαβ Πάσκα Εξ ονόματος της Ευρώπης της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Με μεγάλο ενδιαφέρον διάβασα την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή αποφάσεων σε θέματα διαδοχής και την ε, καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου ώστε να αποφεύγονται κάποια προβλήματα ε, στους συγγενείς του θανόντος σε κάποιο άλλο κράτος μέλος. Εάν ε, πρέπει, εάν ισχύει η επιλογή του τόπου κατοικία κάτι που δεν προσδιορίζεται στο κείμενο, κατά την άποψή μου δεν είναι μια καλή ιδέα. Είναι ένα ασαφής ορισμός που σημαίνει ότι διάφορα δικαστήρια σε διάφορα κρατημέλη θα το ερμηνεύσουν με διαφορετικό τρόπο. Για τόσο ευαίσθητο νομικό κείμενο πρέπει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, πιο σαφείς και να επιλέξουμε πιο συγκεκριμένους και σαφείς ορισμούς. Ο Ντίμητρα Στογιάννοφ, εξ ονόματος των μη εγγεγραμμένων, για 1,5 λεπτό. Благодаря, господин председателю. Въпросите с съдебните... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε σχέση με τις αξιώσεις που προβάλλονται δικαστικώς, θεωρούμε ότι το θέμα αυτό είναι ε, πολύ περίπλοκο. Δηλαδή υπάρχουν υποθέσεις οι οποίες δεν μπορούν να κλείσουν εύκολα. Εγώ όταν ε, σπούδαζα είχα να αντιμετωπίσω ένα τέτοιο θέμα στα πλαίσια του αστικού δικαίου. Πρόκειται για έναν περίπλοκο τομέα. Ο συνάδελφος, ο κύριος ε, Λέχνερ, κατάφερε πολλά. Αυτή είναι η κορονίδα της εργασίες του που θα θυμάται και θα θυμόμαστε για πολύ καιρό. Θα ήθελα όμως να σταθώ και σε κάτι άλλο. Κυρία Επίτροπε, είδα ότι η πρόταση νομοθετικού περιεχομένου δεν έχει τύχει γενικότερη αναγνώρισης. Θα ήθελα η Επιτροπή να καταβάλει μια επιπρόσθετη ε, προσπάθεια. Ε, το λόγο έχει ο κύριος Ταντέος Ζεύκα για δύο λεπτά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 E, w istocie το się to mm, zacząć. także to jest też uwaga do e, planistów. a teraz już e, wracając do sprawy otóż proszę państwa ε, κύριε Ζεύκα, συγγνώμη για την διακοπή, αλλά έχουμε πρόβλημα με τη διερμηνία. Κύριε Ζεύκα, συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά έχουμε πρόβλημα με τη διερμηνία. Ε, μπορείτε να, να, να συνεχίσετε. Κύριε Ζεύκα, συνεχίστε να ομιλείτε. Έχετε τώρα μετάφραση από τα πολωνικά. Δεν είναι βέβαιο. Αφήνω κατά μέρος αυτή την παρατήρηση. Start your speech from the beginning, yes,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 θα έπρεπε να είχαμε καλύτερο οργανώσει αυτή τη συζήτηση. Έχουμε καθυστερήσει μία ώρα για να αρχίσουμε τη συζήτηση πάνω σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Δεν είναι κάτι που επιτρέπεται να συμβαίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτό. Κυρίες και κύριοι, κυρία Επίτροπε, μας κατηγορούν συχνά ότι μιλάμε για θέματα που είναι πολύ απόμακρα από τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών. Δυστυχώς αυτό ισχύει διότι συζητούμε συχνά εδώ για θέματα για τα οποία δεν έχουν νομοθετική αρμοδιότητα τα θεσμικά όργανα τα ευρωπαϊκά. Σήμερα όμως μιλάμε για ένα θέμα ιδιαίτερα σημαντικό για τους πολίτες διότι το κείμενο αυτό θα τους χρησιμεύσει για να αντιμετωπίσουν κάποιες καταστάσεις που θα είναι ιδιαίτερα δύσκολες ε, λόγω του θανάτου κάποιου προσφυλούς προσώπου και η ανάγκη να εισέλθουν στο λαβύρινθο των διατάξεων για τα θέματα διαδοχής. Είναι πραγματικά ένας, μια πολύ δύσκολη πορεία την οποία θα υποχρεωθούν να ακολουθήσουν Ευχαριστώ τον κύριο Λέχνερ διότι το κείμενο αυτό θα επιτρέψει σε όλους τους ενδιαφερόμενους να γνωρίσουν νομική ασφάλεια πολύ μεγαλύτερη μέσα, καθώς κινούνται μέσα σε αυτό τον λαβύρινθο των διατάξεων. Η νομοθετική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δεν, χωρίς να αλλάξει τις διατάξεις του εθνικού δικαίου χωρίς να παρεμβεί στο εθνικό δίκαιο μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε διατάξεις που θα διευκολύνουν τη ζωή ε, πολιτών οι οποίοι έχουν περιουσιακά στοιχεία ή κατοικούν σε άλλη χώρα. Το Ευρωπαϊκό Κληρονομητήριο θα διευκρινίσει, θα προσδιορίσει αυτή την κατάσταση, θα διευκρινίσει το καθεστώς που θα ισχύει για την εκτέλεση της Διαθήκης η έκθεση αυτή πάνω στην οποία εργάστηκε για δυόμιση χρόνια με τις, σε συνεργασία με διάφορους ενδιαφερόμενους ο κύριος Λέχνερ ε, προσφέρει μια ουσιαστική προστιθέμενη αξία. Υπάρχουν πάρα πολλά διαφορετικά νομοθετικά συστήματα σε ό,τι αφορά το δίκαιο της διαδοχής που στηρίζονται σε πολύ πολύ παλιές παραδόσεις για τη δουλειά αυτή, για το έργο αυτό χρειάστηκαν ειδικά προσόντα, μεγάλη εξειδίκευση και πρέπει να το υπογραμμίσουμε ακόμα μια φορά την ε, έργο που επετέλεσε ο εισηγητής μας. Επιβλήθηκαν κάποιοι κανόνες για να αποφεύγονται οι συγκρούσεις ανάμεσα σε διάφορες νομοθετικές διατάξεις και κάτι ακόμα πολίτες θα μπορούν να κάνουν χρήση αυτού του νόμου με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ενημερωθεί σωστά. Ευχαριστώ. Παρακαλώ πάρα πολύ να τηρούμε το χρόνο. <clears throat> Επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Εύελιν Ρέγνα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύρια Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριε Εισηγητή. Το θέμα του κληρονομικού δικαίου θα ε, διευκολύνει τη ζωή ε, πολλών πολιτών και θα ε, ρυθμίσει και τα κληρονομητήρια διότι υπάρχουν πολλοί πολίτες οι οποίοι ζουν σε ένα κράτος αλλά έχουν περιουσιακά στοιχείο σε κάποιο άλλο ενώ τώρα θα έχουν μεγαλύτερη νομική ασφάλεια όταν καταρτίζουν τη διαθήκη τους ή ε, τις τελευταίες επιθυμίες τους και φαίνεται ότι τώρα μπόρεσε ότι τώρα ε, εμποδίζεται να ε, υπάρξει μια ενιαία ευρωπαϊκή ρύθμιση διότι η Μεγάλη Βρετανία και η ε, Ιρλανδία έχουν επαναφέρει την clawback ρήτρα και βλέπουμε όμως ότι στα υπόλοιπα κράτη-μέλη υπάρχουν πολλές αρνητικές επιρροές οπότε δεν μπορούμε να μιλήσουμε μόνο για βρετανικό ή ιρλανδικό πρόβλημα διότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί μία κατάσταση όπου θα επιλέγει ο κάθε ενδιαφερόμενος που θα εγκατασταθεί για να διαθέσει την κληρονομιά του. Θα πρέπει η συζήτηση να γίνει με συμμετοχή όλων των κρατών μελών κατά τρόπον ώστε να υπάρξει μια νέα ρύθμιση πράγμα που μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί και υπάρχει ακόμη νομική ασάφεια. Το Συμβούλιο λοιπόν καλείται να ρυθμίσει δύο θέματα τα οποία είναι ακόμη σε κρεμότητα δηλαδή σαφή ρύθμιση της νομοθεσίας σαφή νομική ασφάλεια χωρίς να υπάρχει αύξηση του κόστους και ε, είναι σωστό να ρυθμίσει κανείς τις διασυνοριακές κληρονομιές αλλά δεν θα πρέπει κάποιος ε, να ε, ε, καταφύγει στην Ιρλανδία ή στη Μεγάλη Βρετανία για να λύσει τα προβλήματά του και ο κύριος Λέχνερ θα μπορούσε να μείνει λίγο παραπάνω να μας λύσει αυτά τα προβλήματα που εκκρεμούν ακόμη. για δύο λεπτά. Ε, Debatujemy nad... Ε, ευχαριστώ. Συζητάμε ένα από αυτά τα τα βασικά ζητήματα της οικοδόμησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς μπορεί να ε, στην ουσία να υπηρετήσει ο νόμος τον μέσο πολίτη. Μιλάμε για το κληρονομικό δίκαιο Υπάρχουν άνθρωποι που δεν ε, συσσωρεύουν καμία, δεν έχουν καμία περιουσία κατά τη διάρκεια της ε, ζωής τους. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ε, υπόκεινται σε αυτή την κατηγορία. Πολλοί όμως έχουν περιουσιακά στοιχεία και γι' αυτό το ζήτημα αυτό πρέπει να διευθετηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πρόταση αυτή είναι ιδιαίτερα πλεονεκτική για τους πολίτες, διευκολύνει θέματα αναγνώρισης, αναγνώρισης του νομικού καθεστώτος στο οποίο υπάγεται κανείς. Αυτό το ζήτημα είναι ύψης της σημασίας και θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον κύριο Λέχτνερ για αυτή την εξαιρετική εργασία. Νομίζω ότι έτσι θα βοηθήσουμε ιδιαίτερα τους Ευρωπαίους πολίτες, θα επιλύσουμε θέματα κληρονομικού δικαίου χωρίς και κληρονομικής διαδοχής χωρίς υπέρμετρο γραφειοκρατισμό. και θα επιλύσουμε διαφορές μεταξύ δικαιοδοσιών. για ένα Thank you, Mr. Um, Αυτός ο κανονισμός θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα νέο καθεστώς. Πιστεύω ότι αυτό το ε, κληρονομητήριο θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν ενιαίο ευρωπαϊκό φόρο ιδιοκτησίας. Δεν θέλουμε ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο να δημιουργηθεί κάτι τέτοιο. Η Βρετανική κυβέρνηση ε, ζήτησε ρήτρα αυτοεξαίρεσης και σε θέματα ε, ευρωπαϊκής αρχής πολλές φορές αντιτάσσεται. Αυτό που, που η ρήτρα αυτοεξαίρεσης δεν με εκπλήσει. Αυτό που με εκπλήσει είναι ότι δεν δέχτηκε να μπει σε αυτό το πλαίσιο. Θα πρέπει να δούμε γιατί δεν ακολουθείται αυτή, η αυτός ο δρόμος σύνεσης εκεί που θα μπορούσε να ακολουθηθεί. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Ραφαέλε Μπαλτασάρε, Περντούε Μινούτη. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, 450.000 είναι τα κληρονομητήρια τα οποία ανοίγονται κάθε χρόνο με μεγάλο κύκλο εργασιών. Όμως ε, υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Δεν ξέρει ο πολίτης σε ποιο δίκαιο να αποτανθεί θα πρέπει να προσθέσουμε ότι τα περισσότερα κράτη-μέλη δεν επιτρέπουν στον πολίτη να επιλέξει τη δικαιοδοσία στην οποία θα υπαχθεί. Γι' αυτό μιλάμε για, πολλές φορές για συμβολιογραφικές πράξεις οι οποίες συντάσσονται σε άλλο κράτος από το ε, κράτος όπου αρχικά άνοιξε το κληρονομητήριο. Δεν μιλάμε για ένα απλό νομοθετικό πλαίσιο, μιλάμε για ένα έργο ζωτικής σημασίας που διέπει το κληρονομικό δίκαιο διευρωπαϊκά. Και Βλέπουμε κατά συνέπεια ότι θέματα κληρονομικής διαδοχής είναι ύψης της σημασίας για την οργάνωση της κοινωνίας. Γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνεισέφεραν στην ε, υλοποίηση αυτού του μεγάλου εγχείρηματος και ιδιαίτερα τον κύριο ε, στα πλαίσια αυτής της ε, νομοθετικής διαδικασίας τον ευχαριστώ εξ ονόματος των εκατομμυρίων πολιτών που θα έχουν ένα εργαλείο που θα τους ικανοποιεί μέσα στα πλαίσια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ε, ακολουθεί η κυρία Καταρίνα Νεβεντάλοβα για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι πρέπει να συμφωνήσουμε ότι η πρόταση της Επιτροπής δεν θα επηρεάσει την νομοθεσία σε εθνικό επίπεδο αλλά θα ε, ε, επιτρέψει τη την εφαρμογή διασυνοριακώς του κληρονομικού δικαίου διότι αυτό προσφέρει νομική βεβαιότητα, είναι κείμενο σαφές και κατανοητό και από τους απλούς πολίτες. Ο κατακαιρματισμός της διαδοχής αποφεύγεται διότι ο τόπος ε, μόνιμης συνήθους κατοικίας μπορεί να ισχύσει κάθε αρμόδια αρχή μπορεί να επιλεγεί από τον έναν ενδιαφερόμενο πολίτη με αυτόν τον περιορισμό ότι θα υπάρχει, προστασία, θα υπάρχει προστασία της οικογένειας και των συγγενών και ότι θα αποφευθούν οι καταχρήσεις Βεβαίως όλα τα εμπόδια, όλα τα μειονεκτήματα δεν μπορούν να καταργηθούν αλλά οπωσδήποτε η κατάσταση ε, μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά. Οι πολίτες θα μπορούν να εξασφαλίζουν το σεβασμό των δικαιωμάτων τους με πολύ ευκολότερο τρόπο και οι, οι νομικές αξίες θα ενισχυθούν και θα δημιουργηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο προστιθέμενη αξία. Άλλων εγγεγραμμένων μιλητών κλείνει με την κυρία Σίλβια Αντριάννα Τικάου για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Madam Commissioner. Κυρία Επίτροπε, για να λειτουργήσει η εσωτερική αγορά θα πρέπει να υπάρχει ελεύθερη κυκλοφορία των φυσικών προσώπων που θα μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους μέσα στα πλαίσια της κληρονομικής διαδοχής. Αυτό σημαίνει εφαρμογή όλων των πτυχών του αστικού δικαίου και ιδιαίτερα όσο αφορά την ε, μεταφορά ε, περιουσιακών στοιχείων σε περίπτωση θανάτου. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε ποιος νόμος, ποια δικαιοδοσία μάλλον ισχύει σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής, δηλαδή από τη στιγμή που ανοίγει το κληρονομητήριο μέχρι τη στιγμή που τα περιουσιακά στοιχεία θα βρεθούν στα χέρια του ευεργετηθέντος. Το Ευρωπαϊκό Κληρονομητήριο θα πρέπει να αποτελέσει ένα βασικό έγγραφο για να καταγράφονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία σε περίπτωση θανάτου και θα πρέπει να εγγράφονται οι πάντες με όλα τα στοιχεία έτσι ώστε κάθε κράτος μέλος να διαθέτει το μητρό του για να γνωρίζουμε κατά πόσο έχει καταβληθεί και ο κατάλληλος φόρος. Θα πρέπει λοιπόν να εφαρμοστεί αυτός ο κανονισμός σε όλα τα κράτη-μέλη. Ελπίζουμε η σημερινή κατάσταση να μην διαιωνιστεί, γιατί βλέπουμε ότι η Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία δεν συμμετέχουν. Κυρία Κατσδιάη, δίνω το λόγο στην κυρία Έλενα Μπασέσκου. Ευχαριστώ. Με την έκθεση αυτή φτάνουμε σε διευκρινήσεις έτσι ώστε να ξέρουμε ποια, ποιες είναι οι αρμοδιότητες και η ε, επακριβής οριοθέτηση θεμάτων ε, κληρονομικής διαδοχής. Επίσης, θα αρθεί η γραφειοκρατία μέσα στα πλαίσια του ενιαίου Ευρωπαϊκού Κληρονομητηρίου. Έτσι θα έχουμε καλύτερη διασυνοριακή διακίνηση και ένα κοινωνικό καθεστώς, ένα με συγχωρείτε νομικό καθεστώς, έτσι ώστε να μην υπάρχουν ρήξεις μεταξύ δικαιοδοσιών. Το κληρονομικό δίκαιο είναι ύψης της σημασίας και για τη χώρα μου αλλά πολλές φορές δεν λειτουργεί βέλτιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Αλάγιος Μεζάρος. Köszönöm, elnök úr. Minden uniós polgárnak joga van ahhoz, hogy Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κάθε πολίτης έχει δικαίωμα και να κληρονομήσει και να κληροδοτήσει. Και ε, υπάρχουν πάντοτε ε, και ενδεχομένως προβλήματα διοικητικά και νομικά και με τη νέα ρύθμιση θα υπάρχει πολύ μεγαλύτερη νομική ασφάλεια η οποία θα επιτρέψει να ε, εξασφαλίσει ε, κανείς σε μια πιο ομαλή διαδοχή μέσω του Ευρωπαϊκού Κληρονομητηρίου το οποίο θα διευκολύνει τις νομικές διαδικασίες. Συνήθως χρειάζεται κανείς πάρα πολλά έγγραφα και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί βλέπουμε ότι ε, δεν μπορούν όλα τα έγγραφα αυτά να υπάρχουν σε μία γλώσσα ενώ τώρα πιστεύω πιστεύουμε ότι όλα θα έχουν ρυθμιστεί και εύχομαι κάθε επιτυχία να ακολουθήσει αυτό το εγχείρημα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ας σκεφτούμε πόσο καιρό διήρκησε αυτή η διαδικασία είναι περίεργο πώς χρειάστηκαν να περάσουν όλα αυτά τα χρόνια για να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα εφόσον υπάρχουν πάρα πολλά περιουσιακά στοιχεία και ακίνητα εις την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει κινητικότητα των εργαζομένων εργαζομένων και ε, πολύ περισσότερα διαζύγια από γάμους. Ε, πρέπει λοιπόν να υπάρχει δυνατότητα ε, να μπορεί κανείς να επιλέξει το δίκαιο διαδοχής του και ο πολίτης θα πρέπει σχετικά με τις αλλαγές του νομικού περιβάλλοντος στην Ευρώπη να επιλέξει πιο δίκαιο επιθυμεί και πρέπει πρέπει να του χορηγήσουμε αυτό το δικαίωμα. Σας ευχαριστώ. Η Αντιπρόεδρος κυρία Ρέντινγκ, εξ ονόματος της Επιτροπής. Κυρία Ρέντινγκ. Thank you. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πιστεύω Ευχαριστώ πρόεδρε, επαναλαμβάνει κυρία Ρέντινγκ. Είναι πολύ ευχάριστα νέα αυτά για τους πολίτες της Ευρώπης υπάρχει σημαντικός αριθμός διαδοχών αναέτος διασυνοριακού χαρακτήρα. Περιορίζουμε τη γραφειοκρατία, διευκολύνουμε τους πολίτες, αυτό πρέπει να κάνουμε για να τους επιτρέψουμε να ασκήσουν τα δικαιώματά τους σε ό,τι αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία η συνεργασία ε, αυτή είναι πρώτη διασυνοριακή συνεργασία για την οποία απαιτήθηκε πολύ τεχνική δουλειά και θα χρειαστεί και πολύ χρόνο οι αντιπροσωπείες για να αντιληφθούν τα διάφορα θέματα και τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ νομικών συστημάτων. Σημαντικό μέρος αυτής της δουλειάς ε, ε, εστιάστηκε στο να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας. Ο μελλοντικός κανονισμός είναι ήδη αντικείμενο συμβιβασμού που θα μπορέσουν να δεχθούν η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο διότι θα αποκομίσουν ουσιαστικά ωφέλη οι πολίτες τους. Εν πάση περιπτώσει, έστω και αν αποφασίσαμε επ' αυτού χωρίς τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας θα έχουν πάντα δύο αυτές χώρες τη δυνατότητα να ενταχθούν αργότερα. Σε ό,τι αφορά το θέμα της ενημέρωσης, συμφωνώ απόλυτα με τους βουλευτές ότι είναι σημαντικό μόλις αυτό το νομοθετικό κείμενο αρχίσει να ισχύει να ενημερωθούν οι πολίτες για τα δικαιώματά τους και τις δυνατότητες που τους παρέχονται. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συμβολογράφων έχει μια ειδική, σχεδιάσει μια ειδική ιστοσελίδα με την χρηματική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μια ιστοσελίδα σε 22 γλώσσες για να ενημερωθούν οι πολίτες για το τι θα σημαίνουν για αυτούς οι νέοι κανόνες. Και είναι σημαντικό η οι όλων των συμμετεχόντων κρατών μελών να ενημερωθούν και να έχουν κατόπιν τη δυνατότητα και εκείνοι με τη σειρά τους να ενημερώσουν τους πελάτες τους για τις δυνατότητες που τους προσφέρονται χάρη σε αυτόν τον νέο κανονισμό. Κύριε Λέχνα, αγαπητέ Κούρτ, ε, σε παρακαλώ και τα δικά μου συγχαρητήρια και τις δικές μου So, jetzt, vielen Dank, Präsident. Ja, vielen Dank. Okay, Κύριε Λέχνερ, θα ήθελα να σας συγχαρώ, να σας ευχηθώ. Υγεία και επένδυση της γνώσης και της εμπειρίας σας επαγαθώ της ε, Ευρώπης των πολιτών. Και θεωρώ με αυτόν πάρα πολύ ευτυχή που συνεργάστηκα μαζί σας κατά την προηγούμενη θητεία στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Έχετε το λόγο, κύριε Λέχνα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για τα ευγενικά σας λόγια κατά την αποχώρησή μου ε, σε τέσσερις ημέρες και 150 λεπτά και θα προσπαθήσω ε, για να, ε, μέχρι την τελευταία στιγμή για να μπορέσει να υιοθετηθεί το έργο μου αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τις σημαντικές συμβολές και θέλω να πω στην Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ήταν ένα πολύ βασικό θέμα και χαίρομαι που μπορέσαμε να καταλήξουμε κάπου διότι ε, γι' αυτό το, ε, λόγω της φύσεως ε, των θεμάτων και του αντικειμένου δεν είναι εύκολο να μπορέσει να υπάρχει μια ικανοποιητική λύση. Πάντοτε θα παραμείνουν και ερωτηματικά και προβλήματα και γι' αυτό θέλω εδώ να αναφερθώ σε ορισμένα σχόλια που έγιναν έγιναν και να πω στην ε, κυρία Ρέντνερ ότι υπάρχει μία παρανόηση. Δεν σημαίνει ότι δεν ρυθμίζουμε το clawback. Απλούστατα με το clawback βλέπουμε πώς οι δωρεές εν ζωή θα μπορέσουν να ληφθούν υπόψη σχετικά με τα κληρονομητήρια. Και αυτά ρυθμίζουν όπως το επιθύμησαν οι Βρετανοί και οι Ιρλανδοί συνάδελφοι. Τώρα, εάν υπάρξει τελικά μία διαφορετική λύση, κάτι διαφορετικό και ίσως ένας άλλος συνάδελφος ξέχασε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή Βρετανοί που ζουν στη Γαλλία, στην, ε, στο Βέλγιο που έχουν ακίνητη ιδιοκτησία στις χώρες αυτές όπου εφαρμόζεται κάποιο άλλο δίκαιο και όχι το Βρετανικό. Οπότε καλό θα ήταν καταρχήν ε, να ρυθμίσουμε τα θέματα λαμβάνοντας υπόψη τις εμπειρίες που έχουμε διαπιστώσει διότι θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ίσως διευρυμένης επιλογής εφαρμοστέου δικαίου αλλά αυτό ίσως θα χρειαστεί μία εικοσαετία και αυτή τη στιγμή θα πρέπει να υπάρχουν να μπορούν οι αρχές να γνωρίζουν τι μέλη γενέστε και αυτό αποτελεί μία μεγάλη πρόοδο για τους Ευρωπαίους πολίτες ευχαριστώ τον Πρόεδρο για τα καλά του λόγια ευχαριστώ τους συναδέλφους και τους συναδέλφους ε, συναδέλφους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η συζήτηση περατώθηκε. Η ψηφοφορία θα δεξαρθεί αύριο στις 12.30 το μεσημέρι. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή.